Dear colleagues, we're we are... Συνάδελφοι όλοι γνωρίζουμε Έχουμε, πως έχουμε μείνει λίγο πίσω ε, στην ημερήσια διάταξη, είχαμε πολλά πράγματα, οπότε περνάμε αμέσως στο σημείο 20 που είναι η αναφορά από την αντιπροσωπεία στην Κύπρο. Υπάρχει μια σύντομη παρουσίαση του σχεδίου ε, έκθεσης ε, που έχω συντάξει εγώ γιατί ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Κύπρο ως επικεφαλής αντιπροσωπείας θα ήθελα να πω βεβαίως πως το ζήτημα των αγνοούμενων είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί όλους γνωρίζετε πως ε, το 63 και 64 είχαμε δει ε, συγκρούσεις μεταξύ των κοινοτήτων και βέβαια το 74 είχαμε την ε, τουρκική εισβολή γύρω στα 2.000 άτομα και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι αγνοούνται και η μοίρα τους μέχρι σήμερα είναι άγνωστη. Αυτό σημαίνει βεβαίως ε, πόνο για τις οικογένειές τους ε, και για να προχωρήσει η εκταφή και η ταυτοποίηση των ε, σωρών τους ε, η Επιτροπή Αγνοωμένων ξεκίνησε να λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και πέρσι το Δεκέμβριο μία αντιπροσωπεία μελών της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ταξίδευσε στη Λευκοσία για να πληροφορηθεί τις νεότερες εξελίξεις σε σχέση με το έργο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Πρέπει να αναφέρουμε πως ε, σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου αυτής της Επιτροπής ε, προήλθε από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ως ε, αντιπροσωπεία λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον κύριο Λόντλετ Σίμπορ, σύμβουλο των ειρηνευτικών δυνάμεων στην Κύπρο, μέλη της Επιτροπής ε, Αγνοουμένων και μάθαμε πώς λειτουργεί αυτή η Επιτροπή. Είχαμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Ε, Επισκεφτήκαμε επίση και το ανθρωπολογικό εργαστήριο όπου αναλύονται τα, οι εκταφέντες ε, σωροί πριν σταλούν δείγματα οστών για ανάλυση DNA. Στο θεσμικό επίπεδο συναντηθήκαμε με την Επιτροπή Αγνοουμένων, με βουλευτές, με τον Υπουργό. Συναντηθήκαμε με συγγενείς των αγνοουμένων και από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τώρα, αν κάποιοι βουλευτές θέλουν να προσθέσουν κάτι... Παρακαλώ να το κάνετε, αλλά λίγο σύντομα για να ε, μην έχουμε και μεγαλύτερη καθυστέρηση. Θέλει κάποιο το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Ε, πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει την έκθεση και νομίζω είναι πολύ αντικειμενική. Ιδιαίτερα στην τελευταία σελίδα που βγάζει τα συμπεράσματα και ακριβώς καλείται το CMP να προχωρήσει για να κάνει investigations, να κάνει έρευνα ε, σε όλες τις θεωρητικές περιοχές στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Το θέμα των αγνωμένων είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικών και ω τέτοιο πρέπει να το δούμε. Οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την ε, αντιπροσωπεία των συναδέλφων που επισκέφτηκαν την Κύπρο και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχίσει. Δεν έχω δει δημοσιευμένο όμω το συγκεκριμένο έντυπο και δεν ρωτούμε, έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Δεν το έχουμε πάρει το τελικό έντυπο για να το δούμε. Προσωπικά έχω κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ε, βλέπω ότι έχουν εσωματωθεί και το χαιρετίζω και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ καλά και αντικειμενικά κείμενα που έχω γραφτεί επί του θέματος. Άλλα σχόλια. Αν όχι, βεβαίω. Θα μοιραστεί η έκθεση. Και επιπλέον. Υπάρχει εδώ πέρα και ένα θέμα, ένα σημείο για πληροφόρηση με την πρόσκληση που απευθύναμε στα μέλη της Επιτροπής Αγνοωμένων να έρθουν στην ε, Κύπρο να μιλήσουν στην Επιτροπή μας. Και κατάλαβα πως θα έρθουν στην συνεδρίασή μας στις 19 Ιουνίου. Ωραία, περνάμε στο επόμενο. Ανακοίνωση της Κομισιόν προς το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Κεντρική Τράπεζα, ΟΚΕ και Επιτροπή των Περιφερειών. Μάλιστα. Ε, εδώ πέρα όμως μου λένε πως πρέπει να είναι παρούσα η κυρία Λεμπάιλ από την Κομισιόν. Ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή έπρεπε να είναι εδώ. 4 και 45. Έρχεται, μου λένε. Ήρθε. αυτό είναι συγχρονισμός. Καλώς ήρθατε. Πάνω στην ώρα. Ευχαριστώ που ήρθατε κυρία Μπάιλ. Στόχο έχουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να έχουν αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνη για να συζητήσουμε τον πίνακα βαθμολογίας του 2013 που ορίζει προτεραιότητες, ε, χρόνους διεξαγωγής των διαδικασιών, ε, ποσοστό εκδίκασης, εκρεμούς, εκρεμής υποθέσεις, ε, εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, εκπαίδευση των δικαστικών διαδικασίες. Ας ακούσουμε λοιπόν από την Γενική διεθνή Δικαιοσύνη την κυρία Φρανσουάς Λεμπαρίλ. Και μετά θα συζητήσουμε. Έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Chair, and thank you for... Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο και σας ευχαριστώ που μου δίδετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω αυτά τα πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία από τις πρωτοβουλίες που λάβαμε και μπορούμε με ικανοποίηση και υπερηφάνεια να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων που ελπίζω ότι έχει τη διαθεσή σας είναι ένα νέο εργαλείο που παρουσιάζουμε με στόχο την ε, πρόθεση αποδοτικών συστημάτων δικαιοσύνης. Επιτρέψτε μου να σας πω γιατί είναι σημαντικά τα αποδοτικά συστήματα δικαιοσύνης κατά την απόψή μας. Πρώτα απ' όλα, διότι στα πλαίσια αυτών των συστημάτων μία δίκαια δίκη είναι σε όλα τα συστήματα δικαιοσύνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βάση της δημοκρατίας και προσθέτει στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ομιλούμε για εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, πρέπει να πούμε ότι οι εθνικοί δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν τις αποφάσεις που αφορούν το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και στην πράξη ενεργούν σαν δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν μιλούμε για δικαιοσύνη η οποία είναι συγκεντρωμένη, αν θέλετε, επικεντρωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πιστεύουμε ότι οι εθνικοί δικαστές όντως είναι οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο στοιχείο που θα αναφέρω για να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα είναι διότι στον τομέα της δικαιοσύνης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε το κλίμα αυτό αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι να μπορούμε να έχουμε αποδοτικά, αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης. Αν υπάρχουν αδυναμίες και δυσλειτουργίες, μπορεί ενδεχομένως να θυγεί και το όλο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το σύστημα δικαιοσύνης και χώρες. Επίσης, ένα συμπληρωματικό στοιχείο για το οποίο εξετάσαμε τα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα είναι ότι ένα καλό τέτοιου είδου σύστημα είναι καθοριστικό για τις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται Και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να παράσχουμε ενίσχυση και βοήθεια σε συστήματα τα δικαιοσύνης τα οποία θέλουν να βελτιώσουν κάποια συστήματα στην, ε, ε, και να τα κάνουν πιο αποδοτικά σε κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα και άλλες χώρες. Γι' αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, το οποίο θα επηρεάσει από αποφάσεις που θα πάρουν κάποιοι επενδυτές για να ε, ξέρουν ότι μπορούν να στηριχθούν σε τέτοιου είδους σωστά συστήματα δικαιοσύνης. Επίσης, το θέμα της ανεξαρτησίας τους είναι πολύ σημαντικό. Εξετάζουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ανεξαρτησία, επαναλαμβάνω, δεδομένου ότι και πάλι πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει αυτούς που θέλουν να πάρουν αποφάσεις να τις πάρουν και με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο όλα αυτά μεταφράστηκαν στο περίφημο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στις συστάσεις οι οποίες υπευλήθηκαν πέρσι έξι χώρες μέλη στα πλαίσια αυτού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις έρευνες για την ετήσια ανάπτυξη. Κάναμε λοιπόν διάφορες συστάσεις για να βελτιώσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους στους διάφορους τομείς η κάθε χώρα. Δεδομένου, όπως σας λέω, υπάρχει διασύνδεση, σχέση μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικής αποτελεσματικής δικαιοσύνης. Και αυτός, η σχέση που υπάρχει είναι πολύ ισχυρή. Έγινε αυτό για κάποιες χώρες καταρχάς και τώρα επεκτείνεται και στις 27. Αυτό το οποίο κάνουμε εδώ δεν είναι πίνακας βαθμολόγησης των κρατών μελών. Παραθέτουμε στοιχεία, αριθμούς και καταρτίζουμε πίνακες ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα συστήματά τους. Επίσης, επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω κάποια από τα ευρήματα βάσει των κριτηρίων τα οποία θεσπίσαμε και των στοιχείων τα οποία είχαμε στην διάθεσή μας. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα ευρήματά μας. Πρώτα πάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το όγκο των υποθέσεων που φτάνουν στα δικαστήρια για να ξέρουμε πώς θα μετρήσουμε το χρόνο που θα χρειαστεί για να επιληθεί κάθε υπόθεση, για να εκδικαστούν οι διάφορες υποθέσεις. Στο εν τρίτο των κρατών μελών η διάρκεια των διαδικασιών είναι διπλάσια τουλάχιστον από ότι στην πλειονότητα των κρατών μελών. Δεν σημαίνει ε, αυτό ότι χρειάζεται πολύς περισσότερο, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να υπάρξει διεκπαιρέωση της κάθε υπόθεσης. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ε, διαμεσολάβησης. Πολλές φορές αν θέλει κανείς να εκδικαστεί μία ε, υπόθεση γρήγορα θα πρέπει να προστρέξει πολλές φορές σε εξοδικαστικές διαδικασίες για την επίλυση διαφορών. Και βλέπουμε στην έκθεσή μας ότι αν οι περισσότεροι χώρες μέλη έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις μεθόδους εναλλακτικής επίρρησης διαφορών, τη διαμεσολάβηση μεταξύ άλλων, δεν την χρησιμοποιούν παρόλα αυτά οι περισσότερες χώρες. Και ελπίζουμε ότι το μέλλον θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι εναλλακτικές διαδικασίες περισσότερα. Θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούνται ευρύτατα σήμερα. Ένα άλλο έβριμα, ένα άλλο αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι η ανεξαρτησία. Τι εννοούμε όταν λέμε με ανεξαρτησία. Τα δεδομένα τα οποία δίνουμε εδώ είναι διαφορετικά από τα άλλα, τουλάχιστον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι μιλούμε εδώ για την ε, αντίληψη της ανεξαρτησίας. Πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ανεξαρτησία βάσει στοιχείων τα οποία έχουμε από την Παγκόσμια Τράπεζα και σύμφωνα με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε ερωτήθηκαν κάποιες επιχειρήσεις κατά πόσον εμπιστεύονται την ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης. Και εδώ είναι πρώτα απ' όλα θέμα αντίληψης της ανεξαρτησίας. Και αυτό όπως σας είπα είναι πολύ σημαντικό για την απόφαση θα πάρει μια επιχείρηση να επενδύσει χρήματα σε μια χώρα. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την ε, αντίληψη της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων. Υπάρχουν άλλες οι οποίες είναι στα κατώτερα κλιμάκια. Θα βρείτε λοιπόν στην έκθεση και άλλα στοιχεία που αφορούν τον πίνακα αποτελεσμάτων, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν να σας δώσω επιγραμματικά τα κύρια αποτελέσματα των αναλύσεων που κάναμε. Επιτρέψτε μου τώρα να προσθέσω ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων που παρουσιάζουμε είναι ο πρώτος. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ένα εργαλείο τελειοποίησιμο, εξελισσόμενο. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τους τομείς τους οποίους σας ανέφερα. Θα εξεργαστούμε περαιτέρω τους δείκτες και την μεθοδολογία που ακολουθούμε, ώστε να γίνει όλο και πιο έγκυρο και ισχυρό αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιούμε μέσα στο χρόνο, ώστε να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους που πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης. Μία από του, ένας από τους τομείς τους οποίους θα μελετήσουμε είναι, επαναλαμβάνω, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως προανέφερα, και στην έκθεση αυτή προς το παρόν έχετε μόνο τους ορισμούς της έννοιας, της αντίληψης της ανεξαρτησίας και σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε και με τα δίκτυα δικαστών και των δικαστικών αρχών που τους ενδιαφέρει η εργασία αυτή ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε στη θέση μας συγκρίσιμα δεδομένα και στοιχεία σε εθνικό επίπεδο και θα είμαστε σε θέση τα επόμενα χρόνια να παρουσιάσουμε πιο πλούσιους συνδυασμούς στοιχείων από αυτά τα οποία έχουμε σήμερα και προέρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Συμπερασματικά. Τι θα γίνει με αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων. Θα αποτελέσει τη βάση των συστάσεων που θα υποβάλουμε στα κράτη-μέλη, αν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο, στα πλαίσια των ειδικών συστάσεων που θα κάνουμε σε κάποιες χώρες. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε είναι να δούμε να καταλήξει σε πρακτικά αποτελέσματα αυτός ο πίνακας και αυτοί οι δείκτες αποτελεσμάτες. Όχι δηλαδή να μας δώσει μόνο κάποιες ενδείξεις του πώς έχουν τα πράγματα, αλλά να βοηθήσουμε τις χώρες, εάν υπάρχει κάποιο στο σύστημα δικαιοσύνης που μπορεί να βελτιωθεί, να βελτιωθεί. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρώτο βήμα. Θα συζητήσουμε την όλη πολιτική ε, των συστημάτων δικαιωμάτων, Θα το μελετήσουμε στην πρώτη γενική ε, συνάντηση που θα κάνουμε που ονομάζεται στα γαλλικά Assis de la Justice, όπου θα έχουμε όλους τους νομομαθείς εκπροσώπους δικαστικών αργών, ελπίζουμε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζουν ότι θα μπορέσετε κι εσείς να είστε παρόντες σε μια συνάντηση στην οποία θα συζητήσουμε τα διάφορα δικαστικά συστήματα και πάλι τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δικαιοσύνη ως συντελεστής ανάπτυξης. Κατά την άποψή μας, πρόκειται για κάτι το απαραίτητο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό τον τομέα της δικαιοσύνης και να τον βελτιώσουμε. Ο πίνακας αποτελεσμάτων, κατά την άποψή μα είναι μια, ένα καλό σημείο κίνηση. είναι μια πρώτη αρχή και θα μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια, ώστε να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και εμείς και τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμπάγιο. Η κυρία Μπάουερ θα ξεκινήσει τη σειρά των σχολείων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για, τα, ε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Και φαντάζομαι ότι δεν ήταν ε, όλοι ικανοποιημένοι και ευτυχεί, μάλλον με τα αποτελέσματα αυτά στις χώρες μέλη και στα αντίστοιχα Υπουργεία Δικαιοσύνης. Τώρα, όσον αφορά τα συμπεράσματα, δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Φυσικά είναι σημαντικό να γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά. Να υπάρχει ένα βήμα συζήτησης, αλλά φοβούμαι ότι αυτό δεν αρκεί. Πολύ θετικό επίσης που θα οργανώσετε αυτή τη ε, διάσκεψη όλων των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών, αλλά ούτε αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτως ε, αρκετό. Επομένως η ερώτηση που προκύπτει είναι τι μπορούμε και εμείς και εσείς να κάνουμε με τα αποτελέσματα αυτά. Ίσως καλό θα ήταν ε, access to justice. Ε, ίσως καλό θα ήταν ε, να καταλάβουμε εάν και η Γαλλία και άλλες χώρες ενδεχομένως ε, μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο με τα αποτελέσματα αυτά. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Ξέρετε, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων των δικαστών, των δικαστηρίων γενικά. Έρχεται πολύ νωρίς. Γιατί ε, όλο το δικαστικό σύστημα διαπιστώνουμε ότι έχει ευρέως διαβρωθεί από την ε, διαφθορά. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων ούτε μπορούμε εκ των υστέρων να επιβάλλουμε κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τι. Θα ήθελα να ακούσω και από εσά ποια είναι η άποψή σας, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, νομίζω ότι η πρωτοβουλία που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ καλή έτσι ώστε να δώσει ε, ένα είδος ε, κατευθυντήριας γραμμής ή προσανατολισμού. Είναι γεγονός, αγαπητή κυρία, ότι ε, υπογραμμίσατε την το άτομο, τον πολίτη μέσα σε αυτό το δικαστικό σύστημα, ε, το οποίο είναι αργό, το οποίο ε, ο πολίτης, ο Ευρωπαίος πολίτης αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ βραδύ και ότι δεν υπάρχει επομένως σωστή απονομή δικαιοσύνης. Ε, Από την άλλη πλευρά και οι χώρες θα πρέπει να έχουν ένα ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί άλλωστε, όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε κι εσείς, οι εθνικοί δικαστές είναι και ευρωπαίοι δικαστές και πρέπει και αυτοί να έχουν ε, έναν προσανατολισμό κοινό και ενδεχομένως ένα πιο εναρμονισμένο συγκεκριμένο ε, μοντέλο, ε, το οποίο σίγουρα θα πρέπει να εναρμονίζεται και με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ ε, σημαντική και επομένως πήρα το λόγο στην ουσία για να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζίμπελ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λεμπάη για αυτά τα οποία μας είπε. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και την ευχαριστώ για το ότι έθιξε το ζήτημα της εμπιστοσύνης που έχει δύο πτυχές, δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, αλλά στο πλαίσιο αυτό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, αρχών ε, και κυβερνήσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτυχή συνεργασία, που νομίζω πως είναι πολύ σημαντική. Νομίζω πως με αυτό το νέο μέσο θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια επιτυχία, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κάποια κατεύθυνση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των κρατών μελών με τον πίνακα βαθμολογίας, να μην ε, τα κατηγορούμε μόνο, να δείξουμε που υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, να διδαχτούμε, να υπάρχουν κάποιες ανταλλαγές. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης ε, και βέβαιως και να βρεθούν και οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα τα εφαρμόσουν. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης ε, εάν μήπως παρά το νέο αυτό μέσο υπάρχουν κάποιες σκέψεις έτσι μέσω πρόθεσμα να επεκταθεί ο πίνακας βαθμολογίες και να αναφερθούμε σε θεμελιώδη δικαιώματα στο κράτος δικαίου για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια, αλλά νομίζω πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε. Σας ευχαριστώ, η κυρία Κίνγκα Γκέντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω πραγματικά οι Υπουργοί Δικαιοσύνης να χαρούν με αυτό το μέσο γιατί θα συνεισφέρει στην οικονομική επιτυχία της χώρας τους και για μένα είναι η πρώτη ε, κύρια ανάγνωση, αναγνώριση του ότι η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης είναι σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία της οικονομίας και ακόμη περισσότερο στην ενιαία αγορά και άρα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και βεβαίως αυτός ο πίνακας βαθμολογίας μας δείχνει τις διαφορές αλλά και την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση από πλευράς αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας ε, της δικαιοσύνης. Νομίζω λοιπόν πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε πώς η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται στα κράτη-μέλη, καθώς η διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Θα θέλαμε λοιπόν να χρησιμοποιείται στην ενιαία αγορά όλο και περισσότερο αυτή η λύση και βεβαίως ε, να υπάρχει και ικανοποίηση των εμπλεκόμενων μερών γιατί έτσι ε, βοηθεί, μπορούμε να βοηθήσουμε και την οικονομία. Και επίσης θα ήθελα να μάθω κάποια πράγματα περισσότερα για τα επόμενα βήματα σας ε, τι προγραμματίζετε. Μιλήσατε για ένα εργαλείο το οποίο εξελίσσεται και μιλήσατε για την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αλλά νομίζω πως ευρία ταινία νομίζω το κράτος δικαίου και η κατάσταση σε μια χώρα καθορίζει την ελκυστικότητα μιας χώρας για επενδυτές ε, και έτσι μπορεί και να επηρεάσει και την οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω κάποια περισσότερα πράγματα και είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσουμε την συζήτηση αυτή με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Λατφόρτ. Ναι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μας έχετε δώσει κάποιο αντίγραφο του πίνακα βαθμολογίας εδώ πέρα. Θα το ψάξω. Α, εδώ είναι. Μάλιστα. Υποστηρίζω πλήρως ε, την πρωτοβουλία αυτή παρά το ότι Είχε δεχτεί κάποιες επιθέσεις ε, στο Λονδίνο και θεωρήθηκε πως προσπαθεί εδώ πέρα οι προσπαθούν οι Βρυξέλλες να εφαρπάξουν πάλι ε, αρμοδιότητες και να ανατρέψουν το σύστημα του αγγλικού δικαίου. Οπότε για να σας βρίζουν στο Λονδίνο κάτι καλό θα κάνετε. Αλλά να σοβαρευτούμε τώρα. Είναι νομίζω κάτι το ουσιαστικό, γιατί όπως είπε και η κυρία Γκέντς, δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά η οικονομία και η ενιαία αγορά και να υπάρχει απαραίτητη εμπιστοσύνη χωρίς κράτος δικαίου. Ακόμα και στο Λονδίνο γίνεται αυτό αντιληπτό. Ε, δεν μπορεί να υπάρξει ε, ενιαία αγορά και να στηρίζει κανείς την ενιαία αγορά χωρίς να στηρίζει κάτι τέτοιο το οποίο θα ενθαρρύνει και θα οθήσει γενικώ ε, την όσους δεν έχουν τις υψηλότερες προδιαγραφές να προσπαθήσουν να τις επιτύχουν. Ε, εμένα μου φαίνεται προφανές, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ε, έτσι ρίχνοντας μια ματιά στο έγγραφο, αφορά κυρίως το ζήτημα της αστικής δικαιοσύνης ζητήματα εμπορικού δικαίου κτλ. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά προφανώς ε, στην Επιτροπή μας ε, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα σε διάφορες ε, διαδοχικές εκθέσεις την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάποια σύγκριση και συγκριτική αξιολόγηση και παρακολούθηση των συστημάτων, το τι γίνεται, όπως είπαμε, τις αστικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, την ποινική δικαιοσύνη, δικονομικά ζητήματα κτλ. Οπότε μας παραπέμπουν συνεχώς την δήλωση του Πρόεδρου της Κομισιόν πέρσι, αλλά νομίζω εγώ και η ομάδα μου θα θέλαμε να δούμε κάποια πρόοδο σε αυτό το μέτωπο όταν άκουσα δε την πρώτη φορά πω υπάρχει πίνακα βαθμολογία για τα θέματα δικαιοσύνη. είπα επιτέλου, έβρικα. Αλλά μετά απογοητεύτηκα. Αλλά βεβαίω είναι κάτι το εξαιρετικά πολύτιμο, δεν υπονοώ όπω δεν είναι, αλλά είναι ε, μόνο ένα πρώτο βήμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λεμπάη πότε μπορούμε να περιμένουμε κάτι ανάλογο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αστικών ελευθεριών και όλα τα ζητήματα που επανειλημμένα λέμε στην Επιτροπή μας. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ως ακαδημαϊκή δικηγόρος και ερευνήτρια έχω αξιολογήσει πολύ θετικά την μεθοδολογία αυτής της έρευνας όσον ε, αφορά τις επιδόσεις στον τομέα της δικαιοσύνης στις 27 χώρες, κυρίως τον τρόπο μέτρησης του ε, δικαστικού τομέα, γιατί ξέρετε ότι εδώ για μας στην Ουγγαρία είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό και μάλιστα απειλούμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διαδικασίες του άρθρου 7 σχετικά δηλαδή με την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα. Ε, ε, επομένως θα ήθελα να ξέρω ε, ποια είναι η επιστημονική μέθοδος. Ναι, ζητά κανείς τη γνώμη των εταιριών του της Διεθνούς Τράπεζας λοιπά. Αυτή δηλαδή είναι η αντικειμενική αδέκαστη άποψη ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλάβει ε, πώς ε, μετράτε αυτό το, αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα τελικά έκανα πολύ καλά που ήρθα γιατί κατάλαβα πολύ περισσότερα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ε, είναι γεγονός ότι και στην ε, Ουγγαρία αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν πειρά ομαδών προς τη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να απελευθερωθούμε από την νέα μορφή απεικιοκρατίας που εφαρμόζουν η Διεθνής η Παγκόσμια Τράπεζα και όλοι οι όμιλοι κτλ. Αλλά φαίνεται ότι εσείς θεωρείτε όλα αυτά πάρα πολύ θετικά πράγματα. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, παραθέτω, στόχος ε, ε, είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επιτύχουν ε, καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε τα στοιχεία, μάλλον βάση στοιχείων συγκρισίμων και αντικειμενικών που μπορούν να ισχύουν σε όλες τις χώρες μέλη. Μπορείτε παρακαλώ να με βοηθήσετε να καταλάβω καλύτερα τι εννοείτε, γιατί είναι αν θέλετε μάλλον τόσο αντικειμενικά συγκριτικά στοιχεία, γιατί τα ζητάτε από την Παγκόσμια Τράπεζα ή από διάφορες corporations ε, και από τη στιγμή που βλέπετε να υπάρχουν προβλήματα και στις 27 χώρες, γιατί ε, το δάχτυλο το κουνάτε μόνο στην Ουγγαρία και την απειλείτε ε, την χώρα αυτή με κυρώσεις. Δεν θα μπορούσατε να πάρετε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα από τις 27 χώρες, γιατί λέτε ότι... Μάλλον εδώ βλέπουμε με τα στατιστικά στοιχεία ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων, αν θυμάμαι καλά, ε, συνεδρίασαν και η Επίτροπος ε, Ρέντινγκ ε, καθώς και άλλοι τέσσερι επίτροποι από την Ολλανδία, τη Φιλανδία και κάποιες άλλες χώρες ε, αναφέρθηκαν ε, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια. debate on how to, how to... Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για πίεση μεταξύ ομοτήμων, ε, λέμε, αναφερόμαστε σε σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φτάνουμε ε, σε αυτό τον πίνακα αποτελεσμάτων, τον οποίο εκτιμώ, τον αξιολογώ θετικά, γιατί βεβαίως είναι ένα πρώτο βήμα ε, προς την οδό της διασφάλισης κάποιων στοιχείων ότι δηλαδή οι χώρες αφού γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα τηρήσουν τους κανόνες της Κοπενχάγης και ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε και εργαλεία στα χέρια μας, τρόπους έτσι ώστε ε, αυτοί, αυτές οι πράξεις ε, να είναι υποχρεωτικές. Αλλά δεν πρέπει κάπως και αυτά που λένε και κάνουν οι υπουργοί να ελέγχονται από τον Από τον πίνακα αποτελεσμάτων. Η κυρία Λεμπάη, όχι, όχι. σας είχα, δεν σας είχα στον κατάλογο. Ασχοληθήκατε κυρίως ε, με αστικές υποθέσεις, γιατί σχετίζονται και με την ανάπτυξη. Εγώ θα ήθελα προσωπικά ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αναφέρεστε ε, στην αντίληψη που έχουμε για την δικαιοσύνη και όχι τόσο σε ε, πραγματικά αντικειμενικά στοιχεία και περιστατικά. Νομίζω ότι οι αντικειμενικοί παράγοντες είναι αυτοί που πρέπει ε, να ελεγχθούν, ας πούμε, η μέθοδος με, τον, με την οποία βάσει, ο τρόπος βάσει, βάσει του οποίου ε, ορίζονται, διορίζονται οι δικαστές ή πώς μπορεί κανείς να πάυσει ε, δικαστές, ας πούμε. Ίσως αυτό θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Επίσης, να σας πω ότι ε, στην ε, χώρα μου ας πούμε μέχρι το 1999 ε, δεν, μπορούσε, δεν μπορούσαν οι δικαστές να υποβάλουν αίτημα. Έπρεπε να κάθονται ήρεμα και ωραία να περιμένουν αν θα τους ζητηθεί να γίνουν δικαστές. Από το 2006 και μετά έχουμε αντικειμενικό διορισμό των δικαστών. Ε, επομένως, ε, επίσης πρέπει να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες ε, στη διάρκεια της έφεσης απορρίπτονται συγκριτικά με τις εφέσεις οι οποίες υποβάλλονται. Επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν υπόνοιες δωροδοκίας δικαστών και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Ε, απ' την άλλη πλευρά είναι πιθανό ε, η έλλειψη αντικειμενικότητας ή αδέκας της κρίσης των δικαστών να οφείλεται σε κάποιες ε, πεπιθήσεις τις οποίες προσωπικές που έχει ο δικαστής. Απ' την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι στην περίπτωση των ανακρίσεων, δικαστικών ανακρίσεων, οι δικαστές κινδυνεύουν περισσότερο να κατηγορηθούν για μεροληψία. Ούτε για αυτά αναφέρεται πολλά. Ε, και σε αυτή την περίπτωση ε, όχι γιατί δεν γίνεται καλά η ανάκριση, αλλά γιατί ενδεχομένως τα ευρήματα δεν είναι αυτά τα οποία ε, θα περίμενε κανείς αρχικά. Α, θέλετε κι εσείς τον λόγο. συγχωρείτε, δεν σας είχα στον κατάλογο. Έχετε τον λόγο. Ναι, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στα αγγλικά και η δεύτερη θα γίνει στα ελληνικά. Διάβασα πως ε, οι δείκτες για τον πίνακα βαθμολογίας του 2013 βασίζονται κυρίως στο χρόνο της διαδικασίας, το ποσοστό επίλυσης και τις εκκρεμείς υποθέσεις και στο τέλος, σελίδα 20 λέει πως τα ζητήματα αυτά θα ληφθούν υπόψη για να προετοιμαστούν οι αναλύσεις της κάθε χώρας ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2013 και επίσης θα αποτελέσουν καθητήριες γραμμές για τη δουλειά που γίνεται στα προγράμματα ε, οικονομικής προσαρμογής. Έχω δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ε, σχέση έχει αυτός ο πίνακας βαθμολογίας με τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής των χωρών, και το, το ξέρω γιατί είμαι Κύπρια, η Τρόικα έχει μεγαλύτερο λόγο από τους ερετούς βουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, έχει λόγο στο τι κάνει η Τρόικα. Αλλά στα προγράμματα αυτά η Τρόικα δεν έχει... Ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν δίνει λόγο στο Κοινοβούλιο. Ακολουθούν κάποια μέτρα λιτότητας, αυτά αποτυγχάνουν και έτσι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών. Οπότε θα ήθελα τα δικά σας τα σχόλια. Γιατί δεν ε, έρχεται να δώσει λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Τρόικα γιατί δεν έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα προγράμματα αυτά οικονομική προσαρμογή. Η δεύτερη ερώτηση είναι στα ελληνικά. Είχε στην... Τη Δευτέρα στην Κύπρο είχαν μαζευτεί όλα τα κοινοβούλια των ευρωπαϊκών χωρών και μιλώντας μαζί τους έχουν πει ότι υπάρχει τεράστια απόσταση και έχει χαθεί εμπιστοσύνη των πολιτών και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Ευρωζώνη και προς τους μηχανισμούς και ενώ χαιρετίζω αυτό το εργαλείο, γιατί πράγματι χρειάζεται ομοιομορφία στον τρόπο που λειτουργούν τα δικαστήρια, διαρωτούμε, όταν καταστραφεί η εμπιστοσύνη των πολιτών από λαθασμένε πολιτικέ που ακολουθούνται σε θεσμικά όργανα, θα χτιστεί με το να έχουμε τέτοιου είδου εργαλεία απλά για να ελέγχουμε ποιε χώρε είναι συμβιβάζονται με τι οδηγίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό το εργαλείο θα ξαναχτίσει πράγματι την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν χάνεται με λαθασμένε και άδικέ αποφάσει που λαμβάνονται από θεσμικά όργανα. Ορίστε, κύριε Λεμπάιλ. Με την ησυχία σας απαντήστε. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πολύ χρήσιμα. Να ομαδοποιήσω λίγο τις ερωτήσεις. Για την ερώτηση του τι θα κάνουμε με τον πίνακα βαθμολογίας. Δεύτερον, οι περισσότεροι με ρωτήσετε ποιο είναι το επόμενο βήμα και συγκεκριμένα ποιο είναι το επόμενο βήμα στο θέμα του κράτους δικαίου. Να απαντήσω τι θα κάνουμε με το θέμα ως έχει. Σημαντικό είναι να αντιληφθούμε πως αυτό το οποίο κάνουμε πρώτα απ' όλα με αυτό το πίνακα βαθμολογίας είναι να συγκεντρώνουμε ε, γνώση, εμπειρογνωμοσύνη, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνώση για το πώς λειτουργούν τα συστήματα της δικαιοσύνης ε, και ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε, όπως είπα, κάποια γνώση. Οπότε, για να απαντήσω κυρίες Μπέο και Παπαδοπούλου, το πρώτο το οποίο θα κάνουμε είναι κάποια από αυτά τα ευρήματα να μεταφερθούν στις συστάσεις ε, της κάθε χώρας που πλέον αποτελούν κανόνα κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πέρσι λοιπόν είχαμε συστάσεις για έξι κράτη-μέλη και τους λέγαμε πράγματα όπως ε, εάν ε, έχουν συστήματα εναλλακτική επίλυσης διαφορών και τα λοιπά. Οι λοιπόν αφορούν το κάθε κράτος μέλος. Διαφέρουν από χώρα σε χώρα και γίνονται εάν απαιτείται. Δεν θα κάνουμε συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχει άμεσος αντίκτυπος των, ε, της γνώσης αυτής ε, στις συστάσεις ε, που κάνουμε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αμέσως υπάρχει μια χρήση και αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό. Δεύτερον, τι άλλο θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Βλέπετε πως για κάποια κράτη-μέλη δεν έχουμε δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει πως τα κράτη-μέλη δεν έχουν καθόλου δεδομένα ή δεν μας τα δίνουν αλλά δεν υπάρχουν ε, τη συγκεκριμένη μορφή. Και οπωσδήποτε θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να συμπληρώσουμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Τι θα κάνουμε μετά λοιπόν. Είναι θα έλεγα ένα εργαλείο το οποίο εξελίσσεται συνεχώς και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι σταδιακά να διευρύνουμε τους δείκτες που έχουμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα οποία είπατε αρκετά από δηλαδή ε, να καταλήξουμε σε κάποια πιο συγκεκριμένα κριτήρια για την δικαιοσύνη. Γιατί δικαίως μιλήσετε για την αντίληψη της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ναι, και αυτό κάνουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και αυτή τη στιγμή τα μόνα δεδομένα που υπάρχουν είναι αυτά της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, ε, για την κυρία Μόβαη. Ε, ζητάμε, ρωτάμε εταιρείε με βάση αυτά τα οποία ξέρετε για αυτές τις χώρες θα επενδύατε σε αυτές. Και είναι μια αρκετά ενδεικτική απάντηση ε, από πλευράς δηλαδή αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Εάν οι εταιρείε δεν θέλουν να επενδύσουν για αυτό το λόγο σε μια χώρα, κάτι λέει αυτό. Οπότε οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τα στοιχεία που έχουμε και αυτός είναι ο λόγος ε, για τον οποίο θα εμπλέξουμε και το δίκτυο δικαστών, τις ε, δικαστικές αρχές στον επόμενο πίνακα βαθμολογίας και έχουν οπωσδήποτε ε, λόγο εδώ πέρα. Επίση, ε, ένα από τα κριτήρια ανεξαρτησίας είναι ο τρόπος διορισμού των δικαστών, ο τρόπος απόλυσης των δικαστών κτλ. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία σε κάποια φάση θα μπουν στο σύστημα αυτό. Δεν σημαίνει πως ε, θέλουμε το ίδιο δικαστικό σύστημα παντού. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν σκοπεύουμε, όπως είπατε, να υφαρπάξουμε αρμοδιότητες και να επεκτείνουμε την αυτοκρατορία μας. Απλά θέλουμε να έχουμε κάποιους δείκτες για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Αλλά βεβαίως ε, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα κράτους ε, δικαίου που έθεσαν αρκετοί από σας και σωστά αναφέρατε με αυτά τα οποία είπε η Αντιπρόεδρος ε, κυρία Ρέντινγκ αυτή την εβδομάδα και τις επιστολές των τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών. Η απάντησή μου σε αυτό είναι πως ο πίνακας βαθμολογίας είναι ένα στοιχείο του κράτους δικαίου. Δεν είναι όλα τα στοιχεία. Συνεισφέρουμε λοιπόν σε αυτή την ανάλυση του κράτους δικαίου και όλοι βεβαίω ε, δεχόμαστε και το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος Μπαρόζο πως ε, δεν υπάρχει κάτι μεταξύ πολιτικής πίεσης και του άρθρου 7 και είναι ξεκάθαρο από τον πίνακα αυτοβαθμολογίας και από τις συζητήσεις που είχαμε σε κάποια κράτη-μέλη πως υπάρχει η ανάγκη να ε, υπάρξει κάτι μεταξύ της ατομικής βόμβας του άρθρου 7 και της πολιτικής πίεσης και οπωσδήποτε θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν είναι κάτι το απλό. Είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει αλλαγή της ε, συνθήκης, μερική αλλαγή τουλάχιστον και οπωσδήποτε πάμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση και ο πίνακας αυτός βαθμολογίας ε, είναι μόνο ένα στοιχείο αυτής της ανάλυσης του κράτου δικαίου. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε, ανέφερε κυρία Μπόιλ την ε, διαφθορά, να έχουμε κατά νου πως τουλάχιστον για δύο κράτη-μέλη έχουμε τον μηχανισμό CDM για να ελέγξει με... στη Βουλγαρία και στη Ρωμανία πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γεγονός είναι πως έχουμε ε, συστήματα για την ε, ε, προενταξιακή πορεία των κρατών μελών και για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν έχουμε κάτι. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με το μηχανισμό αυτό για το κράτος δικαίου που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε αυτό το δίλημα της Κοπενχάγης δηλαδή ότι ε, όλα αυτά γίνονται πρώτη ένταξη και μετά δεν υπάρχει κανένα τρόπο να ελέγξουμε. Εν ολίγης, λοιπόν, ο πίνακας βαθμολογίας είναι ένα πρώτο βήμα, είναι μέρος της ανάλυσης του τι μπορούμε να κάνουμε για το κράτος δικαίου, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί από άλλα μέσα για να εγγυηθούμε το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank Ευχαριστούμε κυρία Λεμπάγια, για τον χρόνο και την ε, ενέργεια που δαπανίστηκε για να μας εξηγήσετε αυτό το σημαντικό εργασίο ανάλυσης και βελτίωσης του συστήματος δικαιοσύνης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσετε και για την ε, προθυμία σας να ανταλλάξουμε από Τελείωσε η σημερινή συνεδρίαση αύριο το πρωί στις 9.